darf sie bitten platz zu nehmen meine damen und herren! καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Τσεχικής Δημοκρατίας σας καλώς ορίζω. Κύριε Ζέμαν, είναι μεγάλη τιμή να σας καλωσορίζουμε εδώ σήμερα. Αναλάβετε το αξίωμά σας με έναν στόχο. Τον στόχο να ενισχύσετε την ευρωπαϊκή πορεία της τσεχικής δημοκρατίας και να ξαναφέρετε τη χώρα στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό σας αξίζει μια μεγάλη αναγνώριση και αναμένουμε βεβαίως την ομιλία σας. Έχει τον λόγο. Mr. President, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κάθε πολιτικό που έρχεται να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει έμεσα ή ρητά το ευρωπαϊκό του όνειρο. Και εγώ θα ακολουθήσω αυτή την χρηστή παράδοση. Πρώτα πρώτα όμως, θα ήθελα να σας αναφέρω τι δεν είναι ευρωπαϊκό μου όνειρο. Εμπνεύστηκα από έναν ε, πασίγνωστο φιλόσοφο τον Λέσσα Κολακόφσκι, ο οποίος είχε δώσει μια διάλεξη που είχε τον τίτλο «Τι είναι ο σοσιαλισμός». Νομίζω το 1957 άρχισε τον ομιλία του λέγοντα. Σύντροφοι, μου ζήτησαν να σα πω τι είναι σοσιαλισμό. Πολύ ωραία. Όμω, πρώτα-πρώτα, να σα πω τι δεν είναι σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμό σύντροφοι, δεν είναι η δολοφονία πολυγών αντιπάλων. Τα σπουδαπέδα συγκέντρωσες δεν είναι η πολιτική κρατούμενη. Δεν είναι η λογοκρισία. Και με αυτό το ύφος συνέχισε για πάνω από μισή ώρα. Εγώ θα είμαι συντομότερος. Σε πέντε λεπτά θα σας αναφέρω τι δεν είναι το ευρωπαϊκό μου όραμα. Πρέπει όμως να προσθέσω ότι στο τέλος της διάλεξής του ο Λέσακ Κόρασεκ είπε και τώρα συνάδελφοι θα σας πω τι είναι σοσιαλισμός. Σύντροφοι. Σοσιαλισμός είναι κάτι το καλό. Αυτό ήταν εδώ. Οπότε να σας πω και εγώ το ευρωπαϊκό μου όνειρο δεν περιλαμβάνει αυτή την ένα η παραλογή μετακίνηση του Στρασβούργου από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο και πίσω. Το όνειρό μου δεν καλύπτει κάποιες βλακίες που περιέχουν κάποιες οδηγίες όπως Φερρυπίν η οδηγία για τους οικολογικούς ε, ελαφρούς λαμπτήρες. Να σας πω επομένως την προσωπική μου εμπειρία ότι το δικό μου όνειρο δεν περιέχει αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική των Βρυξελών, που πολλές φορές δίνει την ε, εντύπωση ενός άμορφου κουτιού. Δεν περιέχει αυτό το επίκεντρο, αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. στο κτίριο που στεγάζεται. Αυτό το άμορφο κακόγουστο κατασκεύασμα. Αυτό ε, ήθελα να σας πω. Το Ευρωπαϊκό τι δεν περιέχει, τώρα να σας πω τι περιέχει. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από κάτι που έχει πει κάποιος άλλος φιλόσοφος. Τσέχος, ο Βάστροφ Γελογκόρσκι Ανέφερε Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη είναι μια πολιτιστική επιλογή. Συμφωνώ μαζί του. Όλοι κάπου γεννηθήκαμε και αυτό δεν το κατακτήσαμε, δεν ήταν η επιλογή μας όμως το να ανήκουμε στην Ευρώπη, το να είμαστε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο προέρχεται από την ελεύθερη μας βούληση. Και αυτό ωφελεί ιδιαίτερα σε περίπλοκες δύσκολες καταστάσεις όπως τώρα. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Πρώτα πρώτα. Πολιτιστικό είναι κάτι παραπάνω από οικονομικό υπολογισμό που υπολογίζει τα κέρδη και τις ζημίες. πολιτιστικό χαρακτηριστικό είναι ένα άθροισμα κανόνων συμπεριφοράς. Και σε μια διαδικασία ολοκλήρωση αυτό το οποίο απαιτείται είναι κανείς να αρχίσει από κάποιους κοινού κανόνες, κανόνες ίδιους για όλους και όχι με ισοπαίδωση όλων. Υπάρχει μια διαφορά. Οι κοινοί κανόνες, Φερρυπίν, είναι η σχέση μεταξύ ελαχίστου μισθού και μέσου μισθού. Όμως ο μισθός, η αμοιβή εξαρτάται από την παραγωγικότητα της εργασίας. Δεν επιδέχεται επομένω ε, ισοπεδά αυτή η κατάσταση, οπότε θα πρέπει εδώ να διέπεται αυτή η κατάσταση από κοινέ αρχέ. Και χρειάζονται επομένω σε πάρα πολλού τομεί τη ευρωπαϊκή πολιτική ε, χρειάζονται αυτοί οι κοινοί κανόνες. Να ξεκινήσουμε με την εξωτερική πολιτική. Ακόμα ισχύει αυτό το ειρηνικό που είχε πει ο ε, Χένρι Τι νούμερο τηλέφωνο έχει η Ευρώπη. Γιατί ακόμα δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική στην Ευρώπη. Και όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε soft policy, ε, ενδοτική, ε, μη υποχρεωτική πολιτική. Σας παραπέμπω στη δεκαετία του 30 τη γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι αυτή η soft policy, χρειάζεται μια κοινή πολιτική. Έχουμε 28 στρατούς. Δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. και ένα μεγάλο όνειρο μακρόπνο είναι ο κοινοστατός, κάτι το οποίο θα ήταν πιο οικονομικό και πιο αποτελεσματικό. Χρειάζεται επίσης εναρμόνιση των φορολογικών πολιτικών μας. Με μεγάλη μου χαρά σας αναγγέλω ότι η Τσεχική Δημοκρατία αναδέχθηκε το σύνολο τη δέσμη μέτρων για τα φορολογικά. Και έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε ισχυρότερη Ευρώπη. Αυτό βλέπω στον οριζόντα. Το συντομότερο δυνατό γιατί εκείνοι οι οποίοι επικρίνουν το ευρώ το οποίο αυτό βλέπουμε στην ορίζοντα για τη χώρα μας είναι αυτοί που φοβούνται το άγνωστο λένε αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό το κύριο είναι σταθεροποιητικός παράγον για την οικονομική ανάπτυξη. Όμως, Ακόμη περισσότερο χρειαζόμαστε κοινού αγώνες στην κοινωνική μας πολιτική. Ξεκινάμε από τον κοινωνικό χάρτη. Χρειάζονται κοινοί κανόνες και στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Και βέβαια χρειάζεται το θάρρος ενός πάρα πολύ σημαντικού έργου και προγράμματος όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτοκινητοδρόμους, ε, πλωτές εσωτερικές οδούς, εσωτερικά ύδατα και θα πρέπει αυτό να είναι κάτι πιο μακρόχρονο από τις τετραετές θητείες. Είναι κατακλείδη συνάδελφοι. Θέλω κάτι να το πω, κάτι υποτύπων παραπώνου και διαμαρτυρίας. Ο κύριος Κονμπεντίτ δεν ξέρω βρίσκεται στην αίθουσα. Όχι δυστυχώς από ό,τι φαίνεται. Προέβη σε μια δήλωση ή διακήρυξη το ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι ενωμένοι οι νέοι Ευρωπαίοι. Εγώ διαμαρτύρομαι γιατί είμαι γέρος Ευρωπαίος, ηλικιωμένος. Αυτό αποτελεί δυσμενή διάκριση επί τη βάση της ηλικίας, κάτι το οποίο είναι κατάφορα ε, αντίθετο στις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν αυτού, τι θα πει να είναι ενωμένοι, τι θα πει ενωθείτε οι Ευρωπαίοι. Αν αυτό σημαίνει κοινού κανόνες, συμφωνώ. Εάν θα πει κάτι που έχει να κάνει με ενοποίηση, είμαι αντίθετος, κάθετα αντίθετος γιατί η ενοποίηση αλλά όπως, και η στολή είναι κάτι το βαρετό, κάτι το γκρίζο και εγώ είμαι κατά ενός κοινού ευρωπαϊκού τυριού, κοινή ευρωπαϊκή μπύρα. Οπότε δεν μπορώ τώρα παρά να σα συστήσω την ε, τσέχικη μπύρα, την καλύτερη στον κόσμο. Πάντω, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ολοκλήρωση. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Όχι ενιαίο ευρωπαϊκό κράτος. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάτι άλλο να σας πω. Από... Το είπε ο για βαθιά μέσα από την καρδιά μου πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το καλό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. By the way, I spoke English in order to reduce your expenses for interpreters and for translation. Yes. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das über das Mikrofon verstehen konnte. Ξέρω αν το καταλάβατε. Ο κύριος Πρόεδρος είπε ότι μίλησε αγγλικά για να κάνει οικονομία στη Διερμηνία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω πως από εδώ πάνω σπανίως έχω ακούσει λόγο που έχει τόσα διαφορετικά μηνύματα και ικανοποίησε όλες τις πτέρυγες της αίθουσας. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη θαυμάσια ομιλία σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Χρειαζόμαστε την Τσεχική Δημοκρατία, μια πολύ σημαντική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι κρίσιμη χώρα και ξέρουμε τώρα πως είναι φιλοευρωπαϊκή. Το αν είναι τώρα η τσέχικη μπύρα η καλύτερη ε, είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε αναλυτικά οπωσδήποτε στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε.